διαδικασίες βάρση του άρθρου 78 του κανονισμού του Κοινοβουλίου. Οι τίτλοι των πράξεων αυτών θα δημοσιευτούν στα πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης. Βάση